Συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Και θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο εξή ότι γίνεται, ε, μπορούν να μας παρακολουθήσουν από το διαδίκτυο. Το σχέδιο ημερήσιας ε, διάταξης έχει διανεμηθεί στις, 13, ε, στις 30 Ιουνίου 2011. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Καζίνη, ο οποίος μαζί με τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στη συνάντηση της ΚΟΖΑΚ, των Προέδρων της ΚΟΖΑΚ στη Βαρσοβία. Γι' αυτό υποθέτω ότι ο κύριος Καζίνη θα βρίσκεται εδώ αύριο το πρωί μπορώ να σας πω ότι την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε μια πολύ καλή συνεδρίαση σε σχέση με τη συνάντηση της ΚΟΖΑΚ. Έχουμε τρία θέματα υπό συζήτηση της κυρίας την έκθεση παρόλο ε, που προερχόμαστε από την ίδια περιοχή είναι πολύ δύσκολο να προφέρω την, ε, το όνομά της, γι' αυτό θα την αποκαλώ Σουζάνα σε σχέση με την ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας μετά την έκθεση Μάρτιν ε, σε σχέση με το δικαίωμα έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια έχουμε τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 του συντάκτη Σαοντάργας. Αύριο το πρωί από τις 9 μέχρι τις 10 έχουμε την συνάντηση των, της συνεδρίας των συντονιστών. Άρα στις 10 θα αρχίσει η συνεδρίαση της Επιτροπής με την ψηφοφορία για την ερμηνεία του άρθρου 51, David Martin. Μετά την έκθεση ε, Ραφάλ Τρασκόφσκι για τις μονομερείς δηλώσεις και ίσως την ερμηνεία του άρθρου 192 που προτείνεται από τον Κάρλο Καζίνη, από τον πρόεδρό μας. Και το τελευταίο θέμα αφορά την ε, γνώμη του Αντιπροέδρου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εάν δεν έχουμε προτάσεις, τροποποίησεις, θεωρώ ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Εάν συμφωνείτε και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε ένα νέο αναπληρωματικό μέλος από τους ε, σοσιαλιστές, μάλλον θα έρθει αργότερα, η Εύελιν Ρέγνερ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο Αντριάν Σεβερίν αποχώρησε από αυτή την ομάδα και έχουμε την Αυστριακή συνάδελφο στη θέση του. Θα ήθελα να εγκρίνουμε τα πρακτικά, σας παρακαλώ, τη συνεδρίαση ε, της 14ης-15ης Ιουνίου του 2011. Νομίζω ότι είναι διαθέσιμα στους φακέλους σας και τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα εάν δεν διαβιβάσετε παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Εάν λοιπόν υπάρχουν παρατηρήσεις, σας παρακαλώ πολύ να τις ε, διαβάσετε πριν από τη λήξη της συνεμερινής συνεδρίασης. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, την ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση η κυρία Μπρόχο ήταν, ε, ορίστηκε μάλλον ε, γονομοδότης για την πρόταση γνωμοδότησης έτσι ώστε να ασχοληθούμε με το θέμα το, της νομικής βάσης για την ηλεκτρονική δημοσίευση. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση όπου η Ευρωπαϊκή Επίτροπη βασίζεται στο άρθρο 352 της Συνθήκης για την ρήτρα ευελιξίας για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ακριβώς προαπαιτείται ομοφωνία και ε, ομόφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Το θέμα αυτό παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και σήμερα θα πρέπει ε, εμείς να αποφανθούμε με βάση τα θεσμικά και διαδικαστικά ε, θέματα που θα αποτελέσουν προηγούμενο δεν γνωρίζουμε ποια διαδικαστικά ε, μέτρα θα ακολουθήσει η Επικεφαλής Επίτροπη. Γι' αυτό θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τη Σουζάνα και θα μπορούσε να μας πει πώς προβλέπει να ασχοληθεί με το θέμα. Μετά θα αρχίσουμε με τη συζήτηση αυτού του θέματος, άρα Σουζάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως είπε ήδη η Πρόεδρος, πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί η ρήτρα, η επωνομαζόμενη ρήτρα της ευελιξίας. Και ήθελα να τονίσω ότι δεν πρόκειται μόνο για το συγκεκριμένο κανονισμό. Συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη πως η επίσημη εφημερίδα των κοινοτήτων πρέπει να δημοσιεύεται επιγραμμικά Οπότε τώρα πραγματευόμαστε τα διαδικαστικά. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να εγκριθεί αυτός ο κανονισμός, διότι η ρήτρα ευελιξίας ακόμη δεν έχει αιτιολογηθεί πλήρως, καθότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση όπου θα εφαρμοστεί αφήστε που στην Τσεχία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται έγκριση από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Συζητήσαμε με τον εισηγητή τη Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και το διαχειριστή administrator. Ούτε και εκείνοι είναι σίγουροι αν επαρκεί η επίσημη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου αν πρέπει να εκπονηθεί μία έκθεση όπου θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί η ρήτρα ευελιξίας. Θα πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχέστερα το θέμα αυτό, διότι θα δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο. Εάν χρειαστεί μόνο ε, επίσημη συγκατάθεση, επίσημη σύμφωνη γνώμη του Ιου Κοινοβουλίου, αυτό σημαίνει ότι για μεγάλες ε, ε, υποθέσεις θα αλλάξει ο τρόπος δημοσίευσης της επίσημης εφημερίδας. Καταλαβαίνετε τις συνέπειες. Επίσης, ζητήσαμε γνωμοδότηση της νομικής ε, υπηρεσίας η οποία απέρριψε τη χρήση του άρθρου 15 ως νομική βάση και ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί. Δεν έχει διασαφινιστεί λοιπόν το ζήτημα. Και πρέπει να συζητήσουμε εδώ δύο θέματα συγκεκριμένα. Θα επιλέξουμε μία εναλλακτική λύση ή θα ζητήσουμε από την Επιτροπή αφετένα ζητήσει διευκρινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση της ρήτρα ευελιξίας, με ποιο τρόπο δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η ρήτρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε το δεύτερο σενάριο, να ζητήσουμε γνωμοδότηση για να αποφύγουμε οποιαδήποτε νομική ασάφεια στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τους ε, συναδέλφους. Έχετε ιδέες, έχετε παρατηρήσεις σχετικά με την ε, ηλεκτρονική δημοσίευση της ε, επίσημης εφημερίδας. Παρακαλώ. Κωνσταντς Δεγκρίπ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο και αν τα φαινόμενα απατούν ότι είναι επίσημο, υποτίθεται τεχνικό και νομικό θέμα, αλλά είναι και ζητήματα ουσίας αυτά που θίγονται σήμερα και τα ανέφερε και η συγγήτριά μας. Και πραγματικό διακύβευμα, δηλαδή η νομική βάση στην οποία ενδεχομένως θα βασίσουμε τον κανονισμό είναι μια νομική βάση που επιφέρει διαδικασία συναπόφασης ή απλής σύμφωνης γνώμης και έγκρισης. Ε, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που διακυβεύεται για το Κοινοβούλιο. Στην πρόταση αυτή, που είναι πάρα πολύ εύστοχη βεβαίως, καταλαβαίνουμε το θέμα αυτό της ηλεκτρονικής έκδοσης ε, της επίσημης εφημερίδας και θα πρέπει να έχει ένα νομικό καθεστώς. Η παρούσα λοιπόν πρόταση, έλεγα, γνωμοδότηση επιλέγει το άρθρο 352 που είναι η περίφημη ρήτρα ευελιξίας. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Είναι αρκετά ευέλικτη όπως λέει το όνομά της η διάταξη αυτή, αλλά το μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι στη απόφαση... αλλά απλώ στην έγκριση του Κοινοβουλίου. Και τώρα ανοίγει η συζήτηση για το κατά πόσο είναι σκόπιμο Euh, euh, και ε, κατά πόσο είναι σωστή η εύστοχη αυτή νομική βάση, υπάρχουν και άλλα ενδεχόμενα και άλλες νομικές βάσεις και άλλα άρθρα της συνθήκης. Το άρθρο 15 ενδεχομένω που αγιάται δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών και ενημέρωσης όλων των πολιτών. Το άρθρο 297 επίσης που ορίζει ότι οι νομοθετικές πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωση δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα. Υπάρχει και άλλο άρθρο 197 το οποίο αφορά την ουσιαστική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου με ανταλλαγή ενημέρωση πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νομική συζήτηση ε, μπορεί να ανάψει πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχει και πολύ υπόβαθρο εκεί και νομικά και πολιτικά ζητήματα προς συζήτηση για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το θέμα και χρειάζεται χρόνο χρειάζεται λέω χρόνο για να ε, μελετήσουμε εις βάθος αυτό το θέμα της ρήτρα ευελιξίας και ε, τις συνέπειές της, το άρθρο 352 όπως είπαμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι μπορεί να μην είναι ίσως το πιο σκόπιμο άρθρο, ε, διότι ακριβώς το να έχει ένα νομικό καθεστώς ηλεκτρονική έκδοση της ε, επίσημης εφημερίδας είναι πολιτικό ζήτημα. Υπάρχει τεράστια δυνατότητα πλέον και του κοινού και των επαγγελματιών και των νομομαθών ε, πρόσβασης και στην νομοθετική μας δουλειά και σε πραγματικό χρόνο με άμεσο τρόπο ηλεκτρονικό. Οπότε είναι ένα θέμα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας ε, στη διαβίβαση των πληροφοριών. Χρειάζεται λοιπόν λίγος χρόνος, όπως σας είπα, για να μπούμε σε λεπτομέρειες και σε βάθος να μελετήσουμε και να είναι περιστατωμένη η νομική ε, γνώμη για το άρθρο 352 ενδεχομένως. Εκ πρώτης όψεως Μπορεί να μην σα φαίνεται τίποτα άλλο αυτονόητο, αλλά υπάρχουν και άλλα άρθρα που σας ανέφερα, 15, 297, 197 και άλλα, που θα μπορούσαν ενδεχομένω να μας χρησιμεύσουν ω νομική βάση. Και για το Κοινοβούλιο, λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και για τις θέσει μεταξύ των θεσμικών οργάνων, τι σχέσει των θεσμικών οργάνων και τι σχέσει μα με του πολίτε. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν αυτό το άρθρο 352 ρήτρα ευελιξίας είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Κωνσταντς. Ο κύριος Χέφνερ ζήτησε το λόγο. Άλλος θα ήθελα να μιλήσει στη συνέχεια, να κάνει κανένα σχόλιο. Μετά τον κύριο Χέφνερ θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας τον κύριο Περιγιώσο. Κύριε Σέφνερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, διότι αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα. Ο Γκέτε, μέγα ποιητή, φιλόσοφο, γερμανό, πολιτικό, είπε ότι το τι ε, πολλές φορές ε, ε, έχει σχέση με το πώς. Δηλαδή, η μέθοδος είναι εκείνη που έχει πολλές φορές σημασία, η διαδικασία, η μεθοδολογία είναι πιο σημαντικότερη καμιά φορά από το περιεχόμενο. Επί της ουσίας δεν έχει κανένας πρόβλημα, όλοι το θεωρούμε σημαντικό. Απλώς εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η νομική βάση γι' αυτό θα πρέπει να είναι το άρθρο 352. Γιατί να επικαλυστούμε τη ρήτρα ευελιξίας. Εγώ θεωρώ το 197 την ε, κατάλληλη νομική βάση που θα περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα και που θα ε, ενισχύει και τη θέση του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μετά από τόσα έχουμε πει μέχρι τώρα, ε, στην Επιτροπή μας, γιατί έκανε αυτό που έκανε που άλλαξε νομική βάση. Και θέλω να ακούσω και τη νομική υπηρεσία. Ε, μελέτησα το κείμενο που μα έστειλε και συμφωνώ απολύτω. Επί της ουσίας συμφωνούμε, αλλά δεν συμφωνούμε τη μέθοδο, το πώ, δηλαδή τη νομική βάση και το άρθρο που προτείνεται με αι. Ε, θα υπερψηφίσω αν επιλεγεί μια πιο λογική ε, νομική βάση. Okay. Thank you very And... Σας ευχαριστούμε κύριε Χέφνερ. Δεν είδα κανέναν άλλον που να ζητάει το λόγο. Ο κύριος Περιός είναι εδώ από την νομική υπηρεσία, όπως σας έλεγα. Οπότε, παρακαλώ, σας ακούμε αν έχετε παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω πως ε, έχει εκδώσει γνωμοδότηση η νομική υπηρεσία προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για αυτό το θέμα. προς το ερώτημα που έθεσε ο πρόεδρος Λένε. Και είναι σχετικά απλό το συμπέρασμα. Είναι μια διαπίστωση. Ποια είναι αυτή. Η επίσημη εφημερίδα που βλέπετε εδώ, σας δείχνω, δημοσιεύεται επί τη βάση μιας απόφασης του Συμβουλίου που χρονολογείται από το 1958 που βασίστηκε τότε στο άρθρο 181 της ε, συνθήκης τότε. Τώρα, έχει αναπαραχθεί αυτούσιο σχεδόν και είναι πλέον το άρθρο 287 ε, της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή είναι η διαπίστωση, πρώτη διαπίστωση νομικής υπηρεσίας. Η δεύτερη διαπίστωση που κάναμε σχετίζεται με τους εφαρμοστικούς όρους του άρθρου 352. Πριν περάσουμε στην εφαρμογή του άρθρου 352, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, πρέπει να τεκμηριώσει ότι ε, οποιαδήποτε άλλη νομική βάση υπάρχει μέσα στη συνθήκη δεν ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για αυτόν τον συγκεκριμένο κανονισμό. Τρίτη διαπίστωση. Μόλις το στοιχειοθετήσουμε αυτό, δεν υφίσταται άλλη πιθανή νομική βάση. αρμόζει να προσδιορίσουμε τους όρους του άρθρου 352 κατά την εφαρμογή του. Δηλαδή, ε, πρέπει να επιδιώκουμε την επίτευξη ενός στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια μιας πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτη διαπίστωση. Η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πληρεί αυτές τις ε, ε, προϋποθέσεις. Δεν μας λέει γιατί το άρθρο 352, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη δυνατή νομική βάση και γιατί η, δημο... η ηλεκτρονική εφημερίδα και η δημοσίευση που βασίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης της Λισαβόνας γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκειμένη περίπτωση ούτως ώστε να θεσπιστεί μια νέα επίσημη εφημερίδα ε, η οποία ε, στα πλαίσια αυτού του κανονισμού θα αντικαταστήσει την ε, επιχάρτου εκδοχή της εφημερίδας, θα την αντικαταστήσει με μια ηλεκτρονική μορφή σε κατεπίγουσες περιπτώσεις βεβαίως. Είναι θέμα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν να διευκρινίσει για ποιους λόγους αυτή η πρόταση για επιγραμμική ε, εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασιστεί στο άρθρο 352 έχοντας πρωτήτερα αποκλείσει όλες τις υπόλοιπες νομικές βάσεις. Ε, στη γνωμοδότησή της η νομική υπηρεσία προφανώς έλαβε υπόψη τις υπόλοιπες νομικές βάσεις ε, ε, που έχουν προταθεί και που αναφέρθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής σας, συγκεκριμένα το άρθρο 15 της ε, Συνθήκης για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, άρθρο 197 ε, ή άρθρο 198. Τελικά, εμείς σταματήσαμε στην πρώτη στάση. Πώς να το πω. Η επίσημη εφημερίδα Ε, βασίζεται στο 191 που είναι το τωρινό 297. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το άρθρο. Να σας πω λίγα πράγματα για αυτό το άρθρο. Εκεί προβλέπεται ότι ε, όλες οι νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το άρθρο αυτό δεν λέει ούτε με ποια πράξη πρέπει να δημιουργηθεί η εφημερίδα, ούτε ποια είναι η ακολουθητέα διαδικασία. Βεβαίως, στην αρχική εκδοχή του άρθρου, που χρονολογείται από το 58, ε, το χάρη σε αυτή την απόφαση το Συμβούλιο ενέκρινε μία γενικού χαρακτήρα απόφαση επί τη βάση μίας ε, διαδικασίας ε, κάπως αλόκοτης. Ε, το Συμβούλιο εφήβρε τρόπον την Α, στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας, δηλαδή της αρμοδιότητας που έχει να λαμβάνει γενικές αποφάσεις. Στα αυτά τα πλαίσια λοιπόν ενέκνε μία ad hoc απόφαση μέσω της οποίας ζητούσε το Συμβούλιο τότε ε, προτάσεις συγκεκριμένες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ύπατη αρχή όπως ονομαζόταν τότε, ε, και απίφθινε την επιστολή, το αίτημα στους πρόεδρους των δύο σωμάτων. Λοιπόν, και πρότεινε το Συμβούλιο να γνωμοδοτεί το Κοινοβούλιο. Φυσικά το Συμβούλιο θα αποφάσισε μόνο του, γιατί αυτό προβλεπόταν τότε στις συνθήκες. Τώρα, Είμαστε εμείς σε θέση να ε, καλύψουμε αυτό το κενό που αφήνει το άρθρο 297 που είναι και η ενδεδειγμένη νομική βάση απαντάει καταφατικά η νομική υπηρεσία διότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας η νομοθετική εξουσία ασκείται από κοινού από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί τη βάση αυτού που θα έπρεπε να είναι η συνήθις νομοθετική διαδικασία. Το λέει εξάλλου μόνο ποια είναι αυτή η συνήθις νομοθετική διαδικασία ή η συναπόφαση. Υπό την επιφύλαξη λοιπόν των διευκρινήσεων που κανονικά θα έπρεπε να δώσει το Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους ε, όρους χρήσης ε, του άρθρου 352, η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το άρθρο 297 που θα συμπληρωθεί από μια διαδικασία που ονομάζεται συνήθις νομοθετική διαδικασία δηλαδή ε, ε, ε, εκείνη η απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει μιας αρχικής πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρε και στη διάθεση ολόκληρης Επιτροπής αν έχετε ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε, μας διαφωτίσατε κάπως επί του θέματος. Χαίρομαι γιατί ο κύριος Χέφνερ είπε ότι ήδη έχει μελετήσει αυτό το έγγραφο. Νομίζω ότι όλοι το έχετε λάβει, δηλαδή τη νομική γνωμοδότηση που προετοίμασε η νομική μας υπηρεσία. Η αποτίμηση της νομικής βάσης αφορά την Επιτροπή Γιούρη δυνάμει του άρθρου 37 αλλά εμείς θα μπορούσαμε να καλέσουμε τη Γιούρη να εξετάσει το θέμα της νομικής βάσης με υπό το φως μάλλον των συζητήσεων της Επιτροπής, δηλαδή θα μπορούσαμε να αποστείλουμε μία ε, επιστολή χωρίς να προδικάσουμε την ε, μελλοντική απόφαση και η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για μια, για μια γνωμοδότηση, όχι ένα απλό σχολιασμό. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ε, ερωτήσεις προς το συνάδελφο. Θα παραμείνει εδώ μαζί μας. Τότε θα ήθελα να κλείσω αυτό το θέμα, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχουν? Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ για τη γνωμοδότησή σας. Νομίζω ότι υπάρχει μια συνένεση, διότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η ρήτρα ευελιξίας αυτό αποτελεί μία βασική αρχή, δηλαδή τουλάχιστον δικαιολογείται από νομικής πλευράς. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας θεωρεί ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία έκθεση, να μας υποβάλει μία έκθεση, διότι η νομική μας υπηρεσία πιστεύει ότι υπάρχουν λόγοι χρήση, ότι οι λόγοι χρήσης της ρήτρας ευελιξίας δεν αρκούν. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Δεν νομίζω. Άρα πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμό 4, που είναι η πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την άσκηση του δικαιώματος έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντικατάσταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής του Απριλίου του 1995. Ελπίζω ο συνάδελφος ο Ντέιβιτ ε, Μάρτιν να επανέλθει. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πω ότι στις 15 Ιουνίου ήδη είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την γνωμοδότηση Μάρτιν. Η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί την απαρχή μιας έκτακτης νομοθετικής διαδικασίας που ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, και έγκρισης μετά από συνένεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αυτή η κατεξαίρεση διαδικασία σημαίνει ότι θα πρέπει το ζήτημα να συζητηθεί σε επίπεδο Επιτροπής πριν εγκρίνουμε το πλαίσιο. Ελπίζω έκτοτε να βρήκατε το χρόνο να εξετάσετε το προσχέδιο του David Martin έτσι ώστε σήμερα να έχουμε μια ιδιαίτερα καρποφόρα συζήτηση. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε συμφωνήσει για μια προθεσμία υποβολής τροπολογιών μέχρι τις 14 δηλαδή Σεπτεμβρίου στις 12 τη νύχτα. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα μπορούσαμε να εξετάσουμε καταρχήν ε, τις τροπολογίες και ο εισηγητής μας θα μπορούσε να επεξεργαστεί ε, τροπολογίες συμβιβασμού που θα υποβάλει για ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 11 Οκτωβρίου. David Martin. Όπως ε, είπατε, είχαμε μία εκτενή συζήτηση επί του θέματος κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Θα Ίσως θα πρέπει να επαναλάβω ορισμένα σημεία αναγκαστικά. Πολλοί συγχέουν τις προσωρινές επιτροπές με τις προσωρινές ερευνητικέ επιτροπές. Πρόκειται για κάτι το εντελώς διαφορετικό. Οι επιτροπές έρευνα σχετίζονται με κακοδιαχείριση, θέματα κακοδιαχείρισης, δηλαδή Πρόκειται για ένα ειδικό νομικό στάτους αυτές οι ειδικές εξεταστικές επιτροπές. Και δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δύο. Είχαμε τρεις προσωρινές εξεταστικές επιστροφές στην Trans BSC και της Equitable Life. Ήταν οι μόνες τρεις προσωρινές εξεταστικές επιτροπές που είχαν συσταθεί. Όπως γνωρίζετε, η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα δυνάμει των κανόνων να ανταποκριθούμε σε αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας και να φτάσουμε σε νέους κανόνες. Βεβαίως αν είμαστε ικανοποιημένοι με τους κανόνες δεν θα προτείναμε τροποποίησεις. Επειδή όμως δεν είμαστε ικανοποιημένοι θα πρέπει να σας να αναφερθώ στα συμπεράσματα της έκθεσης της Equitable Life. Αναφερόταν ότι η Επιτροπή έχει πολύ λίγες εξουσίες, δεν μπορεί να καλέσει ε, μάρτυρες και δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις τη στιγμή που ένας μάρτυρας δεν συνεργαστεί με την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν υπάρχουν κυρώσεις για ψευδομαρτυρία και αν κάποιος δεν ε, έρθει ενώπιον της Επιτροπής. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προσφύγης στα εθνικά δικαστήρια και ε, δεν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν υποβληθούν έγγραφα. Επίσης δεν έχουμε την δυνατότητα να ζητήσουμε τη γνωμοδότηση ενός εθνικού δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της έρευνας. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω σε αυτά τα θέματα, τα συμπεράσματα της ειδική Εξεταστικής Επιτροπής για την Equitable Life. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια τέτοια εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα διοικητικά έγγραφα, τα έγγραφα που κατέχουν φυσικά οι νομικά πρόσωπα, καθώς και κράτος μέλος. Επίσης θα πρέπει οι αξιωματούχοι και οι υπάλληλοι να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε ερωτήσεις. Επίσης θα πρέπει να κλητεύονται μάρτυρες και να έχουμε τη δυνατότητα, να έχουν τη δυνατότητα να εισακουστούν εκεί που κρίνεται αναγκαίο. Και αυτό αφορά την επιλογή μαρτύρων, τη διαδικασία επιλογής μαρτύρων μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας για να μπορέσουν και τα κράτη-μέλη να ορίζουν τους αξιωματήχους. Εάν ζητηθεί λοιπόν μαρτυρία, τότε η Κομισιόν θα αποφασίσει ποιον θα αποστείλει στην ε, Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό ε, μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος είχε άμεση πρόσβαση με τα εν λόγω έγγραφα, τα αμφισβητημένα έγγραφα. Επίσης όμως μπορεί να κρίνουμε ότι αυτό δεν, δεν αρκεί και θα θέλαμε μέσα στα πλαίσια της ιεραρχίας να ακούσουμε άλλους υπαλλήλους και αξιωματούχους που θα κατήχαν πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε την μαρτυρία αυτών των αξιωματούχων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει και η υπηρεσιακή κατάσταση. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να επισυμβεί. Δεν θα ήθελα να το ε, τονίσω υπέρ το δέον, αλλά θεωρώ ότι τη στιγμή που ένας υπάλληλος θεωρεί ότι θα πρέπει να παραβεί το γράμμα του νόμου για να ε, αποκαλύψει πληροφορίες, θα μπορούσε ένας τέτοιος υπάλληλος να γνωμοδοτήσει και να δώσει πληροφορίες σε μια τέτοια εξεταστική επιτροπή. Επίσης, ως προς τις κυρώσεις, μπορούν να ζητηθούν κυρώσεις από μια τέτοια εξεταστική επιτροπή τη στιγμή που ένα πρόσωπο δεν παρέχει έγγραφα, ψευδορκή ή δεν μαρτυρεί ή αν κρίνουμε ότι υπάρχει ε, θέμα δωροδοκίας. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια πραγματική εικόνα των γεγονότων του παρελθόντος. Θα πρέπει να μας ε, δίνουν οι μάρτυρες πραγματιστικά στοιχεία και να έχουμε πλήρη συνεργασία των μαρτύρων αν δεν συνεργαστούν τότε θα ε, ανακύψουν κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές, τις κυρώσεις αυτές δεν μπορεί να τις επιβάλλει η Εξεταστική Επιτροπή, αλλά είτε τα θεσμικά όργανα, είτε εθνικά δικαστήρια ή αρμόδιοι οργανισμοί των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρμοδιότητα και δεν ζητείτε και κάτι τέτοιο να πει δηλαδή η Επιτροπή να αποφανθεί και να πει ότι ο κύριος Χ ε, θα πρέπει να δεχτεί μία κύρωση Χ χιλιάδων ευρώ ή δωροδοκήθηκε οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να εξηχνιάσουμε τα γεγονότα και αυτό με τη συνεργασία των εθνικών αρχών. Αν λοιπόν επιβληθούν κυρώσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες με αυτές που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη. Άρα δεν θα υπερβούμε εθνικά πλαίσια. Και θα πρέπει να δεχτούμε ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να έχει ε, διαφορετικό επίπεδο δικαιοδοσίας, δηλαδή υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ως προς την ιεράρχηση κυρώσεων. Μερικοί συνάδελφοι με ρώτησαν τι γίνεται με αυτή τη διαφοροποίηση κυρώσεων. Υπάρχει αυτό το έγγραφο, το δείχνει ο μιλητής, σε σχέση με τις εξετεστικές επιτροπές μέσα στα πλαίσια των εθνικών συστημάτων δικαιοδοσίας. Υπάρχει αυτό το έγγραφο που μας δείχνει ποιες αρμοδιότητες και εξουσίες υπάρχουν σε κρατικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι πολύ φιλόδοξη αυτή η έκθεση. Και το Κοινοβούλιο εκεί που κρίνει αναγκαίο να συσταθεί μια τέτοια εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να έχει και τις αρμοδιότητες να μπορεί να διεκπαιρεώσει τις εργασίες της. Προτρέχοντας θα μπορούσα να πω ότι δεν θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες να περάσει αυτό το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη όμως με τα άλλα θεσμικά όργανα για να συμφωνήσουμε ως προσαρμοδιότητες. Το 2007 όταν προσαρμόσαμε τους κανόνες, επειδή θεωρήσαμε ότι πρόκειται για αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου, αυτό αμφισβητήθηκε από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, θεωρήθηκε τότε ότι η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να συσταθεί, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω φιλανδικά. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό όταν έχουμε εξεταστικές επιτροπές να έχουν κάποιες εξουσίες και αρμοδιότητες αυτές οι επιτροπές. Ωστόσο, γνωρίζοντας πάντα ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστήριο, είναι νομοθετική εξουσία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη διάκριση των εξουσιών. Άλλο η δικαστική εξουσία, άλλο η νομοθετική και άλλο η εκτελεστική. Όταν εμείς ε, προσάπτουμε σε ορισμένα κράτη ότι έχουν ε, προβεί σε ατασταλίες ή υπάρχουν παρατυπίες, δεν θα πρέπει να ε, υποκαθιστούμε εμείς τη δικαιοσύνη με λίγες εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα. Έχω μια ερώτηση στον εισηγητή. προτείνεται πολλές εξουσίες και αρμοδιότητες για την Εξεταστική Επιτροπή. Μπορούμε να αποτανθούμε και στην Όλαφ και στον διαμεσολαβητή ή σε αντίστοιχα όργανα στα κράτη-μέλη, στους διάφορους συνηγόρους του πολίτη, ας πούμε, ή τις ε, υπηρεσίες δίωξης του οικονομικού εγκλήματος. Θα πρέπει να, να ξέρουμε ε, ποια είναι η εξουσία του Κοινοβουλίου και πού έχουμε εξεταστικέ αρμοδιότητε και πότε. Γι' αυτά θα πρέπει πάντα να τα κάνουμε σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα. Να μην ε, γίνεται διπλή ε, δουλειά και να μην εξετάζουμε διάφορα πράγματα, μάλλον τα ίδια πράγματα σε διάφορα επίπεδα. Επαναλαμβάνω, το Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστήριο. Ε, Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βίλαντ και μετά ο κύριος Χέφνερ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Ε, άλλαξε ο σκιώδης γιατί στην ομάδα μας. Δεν κατάφερα ακόμα να μπω στις λεπτομέρειες. Περάσαν και οι προθεσμίες. Και ε, θα με ενδιέφερε να ακούσω ε, πότε είναι οι νέες προθεσμίες για τις τροπολογίες και τα λοιπά. Θα συζητήσω με τον εισηγητή. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα που μου κάνουν εντύπωση. Δεν θέλω τώρα να σας αναφέρω όλο το εύρος αυτών των θεμάτων με τη σειρά του κειμένου. Καταρχάς, είστε το εξή ερώτημα. Μέχρι τώρα έχουμε ένα κανονισμό και ένα παράρτημα. Πώς είναι αυτά τα δύο σύνδεση μεταξύ τους. Το άρθρο 185 και 186 του κανονισμού έχουν κάποιες διατάξεις πολύ λεπτομερείς ε, και τις έχετε στην έκθεση. Επιπλέον έχουμε και ε, από το 95 το παράρτημα 9 ε, ορισμένα πράγματα που μου φαίνονται πολύ σημαντικά είναι στο παράρτημα και άλλα είναι στο διατακτικό. δεν θα πρέπει να μπουν στα άρθρα όλα τα σημαντικά. Για παράδειγμα, στο άρθρο 2, σημείο 3β, ε, μέχρι τώρα ρύθμιση μόνο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής έχουν πρόσβαση. Δηλαδή όχι ad hoc εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Αυτό για μένα έχει σημασία όταν είναι τα θέματα δύσκολα και ακαθόδη. Ε, επίσης για την προθεσμία άρθρο 2 ε, σημείο 3 ε, γάμα 12 μήνες με δύο φορές ε, δυνατότητα ε, ανανέωσης ή παράτασης ε, ισχύει σήμερα, αλλά καλό θα ήταν στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής να οριστεί, γιατί πολύ καιρό χάνεται στις προκατακτικές ε, εργασίες. Και εγώ θα ήθελα η προθεσμία αρχής να μετράει από την πρώτη συνεδρίαση σύσταση σε σώμα. Και στο άρθρο 3 για την προεκλογική περίοδο, κύριε Μάρτιν, σε θέματα περιβάλλοντος έχω ζήσει κάτι πάρα πολύ λυπηρό. Όταν έχουμε εκλογές ε, μια χρονιά από τον Απρίλιο για να μην πω από τον Μάρτιο δεν μπορεί να πηγαίνει ποτέ αντιπροσωπεία να διαπιστώνει την κατάσταση. Διαφωνώ. Μέχρι ε, τη ε, σύσταση σώμα του νέου κοινοβουλίου θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται η Επιτροπή σε τέτοια δύσκολα θέματα. Ας πούμε με τη ΣΕΒ. θυμάστε τι έγινε με την εγκεφαλοπάθεια. Δεν είναι εκλογικού ενδιαφέροντος το θέμα αυτό. Και το, δηλαδή το Φλεβάρι ή το Μάρτι το 2014 θα αφήσουμε το σφυράκι στην άκρη και δεν θα συνεδριάζει ποτέ η Επιτροπή. Όχι, να συνεδριάσει μέχρι τέλους. Και αν είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα, το νέο κοινοβούλιο μόλις συγκροτηθεί σε σώμα να αποφασίσει νέα εξεταστική επιτροπή χωρίς καμία μετάβαση και χωρίς καμία διακοπή. Αυτή η δυνατότητα τουλάχιστον να προβλέπετε. Κάτι άλλο. Στο άρθρο 5, παράγραφος 2. Δεν θα πρέπει οι μάρτυρες και οι οπειρογνώμονε απαραίτητο να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα ή να, ή να καταθέτουν και κλεισμένων το θυρών. Γιατί αν το γράψουμε έτσι, οποιοδήποτε μάρτυρας μπορεί να έρθει και να λέει θέλω και κλεισμένων το θυρών. Ε, και αυτό θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευκαιρία τη επιτροπή, όχι του μάρτυρα. Στο άρθρο 9. Στα αποτελέσματα των ερευνών δεν βλέπω να λέτε τίποτα για ψήφο μία ψηφία. Θέλω να το γράψετε. Ας πούμε, στο 25% των μελών να υπάρχει δικαίωμα μειοψηφία. Όχι κάθε βουλευτή μεμονωμένα, ξεχωριστά, γιατί αυτό θα ήταν πολύ επιβαρυντικό για τι υπηρεσίε, αλλά το 1 τέταρτο των μελών, όταν έχει άλλη στάση μειοψηφική, να το υποστηρίζουν και οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου και να αντικατοπτρίζεται η άποψη αυτή τη μειοψηφία και στο νομικό κείμενο. Άρθρο 18. Σωστά τονίζεται ότι ε, δεν είναι σε κάθε κράτος μέλος συνήθως να ορκίζονται οι μάρτυρες ε, και δεν είναι και αυτονόητο. Και θα μπορούσα στο 18, στο 2 τουλάχιστον να αναφέρουμε ότι τα κράτη που οι μάρτυρες ορκίζονται στα δικαστήρια ε, να υποχρεώνονται και για τις κυρώσεις ε, να είναι ουσιαστικές, αναλογικέ και αποτρεπτικές, αλλά θα πρέπει να λέμε ότι σε περίπτωση ψευδούς μαρτυρικής κατάθεσης ε, να ε, υφίσταται ο μάρτυρας αντίστοιχα με εκείνα που υφίστατο σε ψευδορκία, σε εθνικό δικαστήριο ή σε εθνική εξεταστική επιτροπή. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και εκείνοι που δεν έχουν καμία τέτοια ρύθμιση ε, εντάξει, να υπόκεινται σε αυτή τη διατύπωση. Οι κυρώσει αυτέ οφείλουν να είναι ουσιαστικέ, αναλογικέ και αποτρεπτικέ. Δύο ακόμα σχόλια. Ένα το ξέχασα, αλλά θα μου έρθει. Ε, στο άρθρο 19. Θα μπορούσα να φανταστώ πάρα πολύ καλά στο σημείο 3 να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει το δικαίωμα να ε, βλέπει τι ε, δυνατότητα υπάρχει ε, μια καταγγελία να έχει και κάποιες επιρροές καθυστερημένες. Αυτό να το καταργούμε. Να πει το Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι η καταγγελία μπορεί να πάει στο δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, οπότε η περίοδος που έπεται της λήξης ε, της περίοδου των 10 εργάσιμων ημερών και τα λοιπά να μην ισχύει. Να του πούμε ότι μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Επίσης, στο παράρτημα, δεν το είδα γιατί δεν το διάβασα. Στο άρθρο 165 παράγραφος 7 έχουμε μια αστεία ρύθμιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει ότι κάθε όργανο θα πρέπει να πληρώνει ε, το κόστος των μαρτύρων. Δηλαδή <laughs> αποφασίζει κάτι ο κανονισμός εις βάρος τρίτων. Δηλαδή όταν κάποιοι άλλοι καλούνται να υπομισθούν κάποιο κόστος, είτε είναι η Κομισιόν, είτε είναι το Δικαστήριο, είτε το Συμβούλιο, είτε τα κράτη-μέλη, τότε ε, θα πρέπει να μπουν αυτά τα θέματα οπωσδήποτε σε αυτό το κείμενο πρωτογενού δικαίου. Αυτά ήταν μια πρώτη ματιά, έτσι. Δεν το έχω μελετήσει το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χέφνερ. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σχετικά σύντομο σε αυτό. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συνάδελφο Μάρτιν για το κείμενό του Σε αυτό το παράδειγμα... Είναι σημαντικά αυτά που λέει τα βασικά ζητήματα και το θεωρώ καλό. Σύμφωνα με τον κύριο Βίλαντ. Θα το συζητήσουμε μεταξύ των σχεδόν εισηγητών σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Από πλευράς μου υπάρχει, είναι δεδομένη και η προθυμία και μπορούμε να δείξουμε πώς δουλεύουν τα κοινοβούλια. Αν θέλουν να δουλέψουν ε, στο Γερμανική Βουλή, ε, πρόσφατα ε, τροποποιήσαμε τα όσα για τις ε, εξεταστικές επιτροπές. Έξι μέλη από έξι πολιτικές ομάδες πήγανε πέντε μέρες σε ένα σημείο συνεδρίασαν πέντε μέρες μόνοι τους και έχει νόημα σε τέτοια θέματα που είναι καθόδη και δύσκολα να αφιερώνουμε και χρόνο θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε η κυρία Μάκη. Βεβαίως και δεν είναι δικαστήριο το κοινοβούλιο. Ούτε το περιμένει κανείς. Ούτε εμείς μπορούμε να δεχόμαστε αγωγές ή μηνύσεις. Ε, στο τέλος μιας εξεταστικής επιτροπής, εξάλλου δεν ε, ε, αποφαινόμαστε, δεν καταδικάζουμε, απλώς διαπιστώνουμε τα πραγματικά περιστατικά. θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να κλητεύουμε μάρτυρες ε, και αναγκαστικά να προσαγάγονται εάν αρνούνται να έρθουν. Γιατί πολύ συχνά μας κοροϊδεύουν, μας εξαπατούν στο κοινοβούλιο και δεν έχουμε τα εργαλεία και τα μέσα εκείνα που να υποχρεώνουν τους ενδιαφερομένους να έρχονται εδώ. Ε, αλλιώς είναι εξεκρέμαστη αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Γι' αυτό τόσο σπάνια τη χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα, γιατί είναι ακριβώς κάτι το οποίο δεν έχει ε, την απαραίτητη πλαισίωση και τις δυνατότητες που χρειάζεται. Ε, είναι λοιπόν καλό το έγγραφο αυτό, βάση για την εργασία. Πολύ καλό και πολύ σημαντικό, το είπε και ο συνάδελφος Βίλαντ, να έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφεται η ψήφος της μειοψηφίας Κατά την εμπειρία μου δεν συμβαίνει πάντα κάτι τέτοιο. Δεν είναι πάντα η πλειοψηφία υπέρ του να διαλευκαθούν τα πάντα. Ε, σε ορισμένες εξεταστικές επιτροπές έχω την εμπειρία ε, ότι μπόρεσαν να διαλευκαθούν κάποια θέματα μόνο επειδή επέμεινε μια μειοψηφία και ενδιαφερόταν και τα προώθησε αυτά τα θέματα. Και έχω και μια ερώτηση προς τον David Μάρτιν. Ε, κατάλαβα εγώ ως εξής τη διαδικασία. Η ιδέα είναι όταν γίνει τριμερής διάλογος, γιατί είναι και έκθεση πρωτοβουλία και πρέπει να πάμε σε τριμερή διάλογο. Εσεί, ω συζητητή τελικά και ο πρόεδρο τη επιτροπής μα, θα κάνετε τι διαπραγματεύσει. Αλλά εγώ κατανοώ τον κανονισμό ω εξή. Θα πρέπει να συμμετέχουν όλε οι πολιτικέ ομάδε στο βαθμό που το επιθυμούν να μπορούν να συμμετέχουν δηλαδή. Ε, για παράδειγμα στον τριμερή διάλογο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών έτσι έγινε ε, και δεν ήταν και κανένα εμπόδιο αυτό, ούτε δυσκόλεψε ε, τη διαπραγμάτευση, μάλλον την υποστήριξη. Είναι σαφέστατο ποιο ε, ηγείται στι διαπραγματεύσει, είναι ο εισηγητή και ο πρόεδρο. Αλλά τώρα να συμμετέχουν, να είναι παρόντε και όλοι εισηγητέ ή συντονιστέ άλλων πολιτικών ομάδων έχει πολύ μεγάλο νόημα και θα παρακαλούσα και θα το προτείνω κιόλα να ισχύσει για αυτόν τον τριμερή διάλογο. Μάλιστα, λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία όταν κάναμε την κοινή μας έκθεση, πραγματικά. Ο κύριος Βίλαντ ξαναζήτησε το λόγο. Ε, μετά κανένα άλλο ο εισηγητή ξανά για να ολοκληρώσει. Ναι. Το θυμήθηκα αυτό που ήθελα να σα πω που μου είχε διαφύγει. Ε, στο έγγραφό του ο εισηγητή, ε, βεβαίω τον οποίο και εγώ ευχαριστώ, λέει ότι η διαδικασία ε, έχει αλλάξει και το Κοινοβούλιο δεν αλλάζει ε, μόνο την προηγούμενη απόφαση, αλλά προτείνει νέο κανονισμό. Ναι, αλλά στο νέο κανονισμό θα πρέπει να ε, είναι ξεκάθαρο ότι η παλιά ρύθμιση καταργείται. Αλλιώς ε, κινδυνεύουμε το παλιό κείμενο να θεωρηθεί ερμηνεία και να το χρησιμοποιούμε και δεν είναι πάντα επιθυμητό κάτι τέτοιο και όχι μόνο σε ερμηνεία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και θα πρέπει να το πούμε κύριε Μάρτιν, ρητά στο νέο κανονισμό, στο παράρτημα 9 συγκεκριμένα, η παράγραφος 5. Για ένα πραγματικό γεγονός που είναι αντικείμενο μιας εξεταστικής επιτροπής, μπορεί μια προσωρινή επιτροπή να συστηθεί μόνο σε περίπτωση που έχουν παρέλθει από την προηγούμενη έκθεση ε, τουλάχιστον 12 μήνες και έχουν, και έχουν εμφανιστεί νέα πραγματικά περιστατικά. Όχι μόνο να έχουν περάσει 12 μήνες, να έχουμε νέα ε, δεδομένα. Αν θέλει κάποιος κάτι τέτοιο, εγώ θεωρώ οπωσδήποτε να παρέλθουν 12 μήνες σωστό, αλλά να υπάρχουν νέα ουσιαστικά και βαριά στοιχεία. Ας πούμε, διαπιστώνεται ότι κάποιος μάρτυρας ε, ψευδομαρτύρησε και μετά έρχεται και μας κατακλίζει ένα σωρός ε, εγγράφων. Δεν μπορεί να περιμένει το Κοινοβούλιο 12 μήνες με σταυρωμένα τα χέρια. Ε, εντάξει, υπάρχουν όρια, τα αναφέρατε, αλλά σε όλα αυτά τα όρια θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση στις εξεταστικές επιτροπές να είναι σκύλος όχι μόνο που να γαυγίζει αλλά και να δαγκώνει. I'm very pleased that uh, you remembered what Καλά που το θυμηθήκατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε. Θα μπορούσε ο εισηγητής ε, να δώσει και εκείνος κάποιες απαντήσεις. Thank you. On, on the last point, which was... Αυτό το τελευταίο πολύ ωραία το είπατε. Περί αυτού πρόκειται. Θέλουμε να μπορεί να δαγκώνει ο σκύλος, όχι μόνο να γαυγίζει. Και αυτό με επαναφέρει σε αυτά που είπε η κυρία Γετεμάκη. Δεν είμαστε δικαστήριο. Από πλευρά διαδικασία αν κάποιο δεν θέλει να συνεργαστεί ή ψευδοκεί κτλ. κτλ. Δεν ε, φέρουμε εμεί ευθύνη για την ε, τιμωρία του, παραπέμπουμε το θέμα στις εθνικές αρχές. Δεν μπλεκόμαστε εμείς ε, στη νομική διαδικασία, αλλά και στα συμπεράσματα μόνο συστάσεις μπορούμε ε, να εκδώσουμε. Δεν έχουν καμία νομική ισχύ ε, θα εφαρμοστούν οι συστάσεις μας ενδεχομένως από τις εθνικές αρχές. Τα, τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής, όποια και αν είναι αυτά, θα εφαρμοστούν ενδεχομένως από τις εθνικές αρχές. Και φυσικά θα συνεργαστούμε με τον διαμεσολαβητή και καλά είπατε ότι το άρθρο 4 ξεκαθαρίζει πως ε, όταν ε, τρέχει μία δίκη, συνεχίζεται μία δίκη, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ε, αν τώρα αρχίσει μία δίκη μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, δεν προτείνουμε να ε, λήξει η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα κρίνει η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή αν είναι ενδεδειγμένο, αν ξεκινήσει νέα δίκη, έτσι. Ε, αν υπάρχει νωρίτερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν τώρα έχει συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή και κατόπιν προκύψει δίκη, τότε στη διακριτική ευχέρεια της Εξεταστικής Επιτροπής να αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι. Άρα προσοχή, δεν θέλουμε να γίνουμε δικαστήριο, δεν είμαστε δικαστήριο, ασχολούμαστε με κακοδιαχείριση ή άλλες παραβιάσεις ε, του, της νομοθεσίας της Ένωσης και διεξαγάγουμε έρευνες. Ο κύριος Βίλαντ έκανε κάποια λεπτομερή σχόλια, δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, ε, θα αναφερθώ πιο πολύ στα γενικά του σχόλια. Δίκιο έχετε ότι πρέπει να ακούγεται και άποψη της μειοψηφίας. Στους συντονιστές κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο. Τι συνιστά μειοψηφία. Ένα άτομο, διάφορα άτομα, πόσοι. Πώς, ε, ποιος αριθμός απαιτείται για να δημοσιευθεί μια έκθεση με την άποψη της μειοψηφία. Επίσης δίκιο έχετε και το εξηγώ μέσα στην αιτιολογική μου έκθεση με σαφήνεια πρόκειται περί νέου κανονισμού. Άρα καταργείται, ακυρώνεται ο παλιός ο κανονισμός με την έγκριση του νέου. Δεν υπάρχει επικάλυψη, δεν ε, μπορεί κάποιος να παραπέμψει στον παλαιό κανονισμό. Αυτό που είπατε για τη λήξη της θητείας. Ναι, είναι η τρέχουσα πρακτική. Όλες οι εργασίες λήγουν με το που λήξει η θητεία. Νομίζω θα ήταν ασύλληπτο να φανταστούμε ότι ιδιαίτερα μια εξεταστική επιτροπή να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ε, εκλογικής αναμέτρησης. Και δεν είναι κάτι που ξαφνικά εμφανίζεται τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, το Μάρτιο, με εξεταστική επιτροπή ε, από το τίποτα, από το πουθενά όπως λέμε, επίτηδες χρησιμοποιώ τον ίδιο όρο μέσα ε, οπότε δεν τίθεται καν τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή αν πριν από τις εκλογές ε, ε, συμβεί κάτι την άνοιξη ας πούμε μου φαίνεται λογικό να αφήσουμε τη συγκρότηση τη Εξεταστική Επιτροπής για, για το νέο κοινοβούλιο όχι να ξεκινήσουμε κάτι που θα πρέπει να σταματήσει Είπατε και διάφορα άλλα τα οποία μεταξύ άλλων έχουμε συζητήσει με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, κύριε Χέφνερ, θα χαρώ πολύ να περάσω χρόνο μαζί σας. Ελπίζω να μην είμαστε και κλεισμένοι για πέντε ολόκληρε ημέρες. Τέλος πάντων, οι σκιώδεις καλό θα ήταν να κάτσουν, να συζητήσουν... Ε, χρειάζεται πάντως η ευρύτερη δυνατή υποστήριξη στο Κοινοβούλιο από το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των πολιτικών ομάδων πραγματικά θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να συμμετάσχουν όλες οι πολιτικές ομάδες ε, στη συζήτηση. Σχόλιο του κυρίου Βίλαντ εκτό μικροφώνου. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι, δεν χρειάζεται. Μπορούσα να προσθέσω κάτι, αλλά δεν χρειάζεται. Μα έχετε χρόνο. Θυμηθείτε όλοι ότι υπάρχει το έτοιμά σας στο άρθρο 20. Ε, ε, η 95-165 επαναλαμβάνεται η απόφαση Τη 19η Απριλίου του 1995, κάτω 167 ευρατών Υπάρχει αυτό ήδη. Σας ευχαριστούμε για τι παρεμβάσει σα και να σας πω και κάτι πάλι, γιατί το είπα πριν, αλλά έφτασαν κάποιοι αργοπορημένοι. Αποφασίσαμε ήδη για την καταληκτική ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα για τις τροπολογίες σας. Η πρώτη εξέταση των τροπολογιών μπορεί να γίνει στην τακτική μας συνεδρία στις 19 Σεπτεμβρίου και κατόπιν ε, ο εισηγητής μπορεί να προετοιμάσει τις συμβαστικές στην Επιτροπή στις 11 Οκτωβρίου στην επόμενη συνεδρίαση. Το επανέλαβα όπως είπα για τους αργοπορημένους. Το πέμπτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 12 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο όλα τα τμήματα. Ο, ε, ο εισηγητής μας, συγγνώμη, ο κύριος Σάνταργκας, είναι εδώ με ε, τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της συνθήκης ε, Λισαβόνας αρχίζει η εφαρμογή του σε βάση της διαδικασίας, ε, κατάρτιση διαδικασίας του προϋπολογισμού και τα σώματα του Κοινοβουλίου, επιτροπέ θα αντιμετωπίζουν περιορισμού και δυσκολίε. Οι δυσκολίε έγκυται αφενό στο ότι όταν συνεδριάζουν οι επιτροπέ τον Ιούλιο, η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού τη Επιτροπή δεν είναι γνωστή. Αφετέρου, υπάρχουν περιορισμοί του δικού μα ημερολογίου και άρα καθίσταται ε, απαραίτητο να προσδιορίσουμε σε επίπεδο επιτροπών και κοινοβουλίου τις ε, προθεσμίες. Ε, δηλαδή, προσδιορίστηκε η ημερομηνία στην 8η Σεπτεμβρίου, που είναι η πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας μετά την καλοκαιρινή διακοπή. Είπαμε ότι δεν θα ήταν... υπάρχουν μικροφωνισμοί η λύση ως στην διαδικασία για την Επιτροπή που προτείνεται είναι η εξής. Ε, σήμερα παρουσιάζεται το σχέδιο και κάποιες τροπολογίες από τον εισηγητή. Ε, υποδεικνύει ποια είναι η θέση του. Αυτά βέβαια υπάρχουν σε μελλοντικές αποφάσεις του Συμβουλίου. Έτσι. Μετά ορίζεται η ε, καταληκτική μερομηνία για τις 29 Ιουλίου το μεσημέρι κατόπιν μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες ε, για την έκθεση του κυρίου Σάντεργκα ε, τα μέλη της Επιτροπής ε, και ισχύει η ίδια καταληκτική ημερομηνία που είπαμε προηγουμένως. Στη συνέχεια θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας συμφώνησε ο Πρόεδρος ναι, να λάβει χώρα αυτή η συνεδρίαση κατά τη μεσημεριανή διακοπή την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου και περιμένουμε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Είναι η εβδομάδα των πολιτικών ομάδων. Από τις 12.30 ε, μέχρι τη 1 και 4 θα συνεδριάσουμε λοιπόν εκτάκτως ε, και θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας ε, που θα εξηγήσει τις προτάσεις του στην Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να πούμε τα εξής. Ως προς τον ε, προπολογισμό, γενικά είμαστε ικανοποιημένοι από τις ε, προτάσεις όπως έχουν διατυπωθεί. Όμως ε, θα πρέπει να πω ότι δεν έχουμε ακόμα την επίσημη θέση του Συμβουλίου επί του θέματος. Έχουμε ορισμένους αποήχους μετά τη συνεδρίαση της Κορεπέρ και οι άλλες επιτροπές θα πρέπει να αναμείνουν την κύρωση των αποφάσεων από το Συμβούλιο. Εμείς δεν θα πρέπει να υποστούμε περικοπές και τουλάχιστον στις γραμμές που μας απασχολούν περισσότερο δεν θα γίνουν σημαντικές περικοπές. Θα ήθελα να πω ότι ασχοληθήκαμε με την ε, χρηματοδότηση των πολιτικών ταμείων, όπου η Επίτροπη προβλέπει μία μικρή αύξηση σε σχέση με το περσινό έτος. Αυτό αντικατοπτρίζει και τη θέση της Επιτροπής μας. Σε σχέση με τις άλλες γραμμές του υπεροπολογισμού, μας απασχολεί εν γέννη το θέμα και έχουμε υποβάλει τις τροπολογίες μας έτσι ώστε οι χρηματοδοτήσεις να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με την περσινή χρονιά. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι μπορούμε να παραμείνουμε στη θέση μας. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τη θέση της Επιτροπής και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα υποστηρίξει τη θέση της Κορεπέρ όπως έχει διατυπωθεί και θα υποβάλει τροπολογίες, τροπολογίες που έχουμε υποβάλει εμείς. Αυτά τα ολίγα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε τον εισηγητή. Υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο, να σχολιάσουν. Ε, αν όχι, τότε να σας πω ότι ο Ενρίκε Γκερέιρο ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Γι' αυτό θα υποβάλω εγώ τα σχόλιά του και θα επανέλθει το Σεπτέμβριο. Ε, ε, Όπως ξέρετε, είχε στο παρελθόν αναφερθεί αυτή η θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου και στα μέσα Ιουνίου έγινε αυτή η διατύπωση. Γι' αυτό θα πρέπει να πω ότι ο προϋπολογισμός του 2012 έχει υποβληθεί σε μία ε, περίοδο χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει πλήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ε, γίνουν περικοπές ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα επιτροπής μας ως προς την ηθαγένεια, ε, ε, τηλεπικοινωνίες, διοικητικά. Έχουν ήδη γίνει περικοπές και δεν θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω περικοπές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χάρηκα διότι τα οι πολιτικές ομάδες και τα κόμματα είπαν ότι θα πρέπει να ισχύσει κάτι τέτοιο. Στην προηγούμενη γνωμοδότησή μας είπαμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην επικοινωνία με τους πολίτες και θα ήθελα να μας υπενθυμίσω ότι το 2012 θα αρχίσουν οι πρωτοβουλίες των πολιτών και τα πολιτικά κόμματα καθώς και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα θα ασχοληθούν με θέματα πρωτοβουλίας, που θα είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Και στο προσχέδιο γνώμης υπάρχουν ορισμένες ιδέες που τόνισε ο Σε σχέση με τη θετική πλευρά υπάρχει ε, μία γραμμή και μία αύξηση για τις πληροφορίες με τα ΜΜΕ ως προς πιστώσεις υποχρεώσεων από αρνητικής πλευράς ως προς εταιρικές ευρωπαϊκές σχέσεις υπάρχει μία φθήνουσα απορία. Η πιστώσεις υποχρεώσεων του 2011 της Europe for Citizens ε, για να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να τύχουν αύξησης, κάτι το οποίο δεν έγινε. Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός για τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών είναι ε, κάτι το οποίο θα έπρεπε να προωθηθεί. Το 2012 όμως δεν υπάρχουν κονδύλια για τις πρωτοβουλίες ε, των πολιτών. Γι' αυτό θα μπορούσαμε και εμείς ως ομάδα να υπογραμμίσουμε ορισμένες πλευρές. Το 2012 υπάρχει μια γραμμή ε, ενός εκατομμύριου ευρώ για τη, τις πρωτοβουλίες των πολιτών για το 2013. Το ίδιο αφορά και το ΜΜΕ και την επικοινωνιακή μας πολιτική. Από αρνητικής πλευράς, οι δαπάνες για τους πολίτες μειώνονται κατά 22,4%. Γι' αυτό η Ευρώπη για τους πολίτες έχει μειωθεί κατά 16.000 ευρώ σε σχέση με την, ε, τα διοικητικά έξοδα υπάρχει μία μείωση 20.000 ευρώ. Είναι πολύ λυπηρές αυτές οι μειώσεις γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ε, online εφαρμογή της ε, επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έκθεση αυτή θα προωθηθεί ήδη από τη Δευτέρα, όπως είπαμε με τη Σουζάνα. Πιστεύουμε ότι η δημοσίευση επί χάρτου θα ισχύσει για ένα μεταβατικό διάστημα σε σχέση με την ηλεκτρονική δημοσίευση. Γιατί μιλάμε για 458.000 ευρώ. Αυτά ήταν τα σχόλια του Ενρίκε Γκερέιρο και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ρωτήσω κατά πόσο κάποιος θα ήθελε να σχολιάσει περαιτέρω το θέμα του προϋπολογισμού. Εάν όχι, εάν υπάρχουν... Α, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, εντάξει. Αυτά. Να σας πληροφορήσω λοιπόν με μεγάλη χαρά ότι αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια θα διακόψουμε τις εργασίες μας και θα τα πούμε αύριο στις 10. Από 9 με 10 έχουμε την συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Ευχαριστεί η Πρόεδρος και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε. Καλό σας απόγευμα και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10.